να ανακληθεί γιατί θα ζημιώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Με αυτή την τελευταία παρέμβαση ε, κλείσαμε αυτό, το ολοκλώσιο αυτό το σημείο ημερήσιας διάταξη. θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά την έκθεση του κυρίου Στέρντι ε, για σχετικά με τους φραγμούς, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Έχει το λόγο ο κύριος Στόρντι για τέσσερα λεπτά. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φέτος το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις και επεσήμανε τη σημασία του να ξεπεραστούν τα εμπόδια στο εμπόριο. Ήταν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μιας ευρείας σειράς μη δεσμολογικών εμποδίων η, πολιτική, στρατηγική της πολιτικής κυρίως επικεντρώνεται στην κατάργηση των δασμών. Όμως η επιμονή αυτών των δαπανηρών ε, εμποδίων στο εμπόριο εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι όλο και περισσότερο οι χώρες χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα προστατευτικά μέσα. Την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος ο Επίτροπος Εμπορίου ε, προειδοποίησε την Επιτροπή μας για το νέο κύμα προστατευτισμού από τους στρατηγικούς μας εταίρους. Το 2020 μπορεί να εκπληρωθεί η εμπορική πολιτική μόνο αν αντιμετωπίσουμε παραγωγικά αυτά τα εμπόδια στο εμπόριο. Η έκθεση αυτή συμβολίζει μια κοινή δέσμευση να προχωρήσουμε με, μια, ε, με θέματα στο θέμα του εμπορίου που θα προκαταλάβει και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Θέλουμε να καταργήσει ή τουλάχιστον να περιορίσει, περιορίσει τα εμπόδια στις δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θέλουν να, έχουν πρόσβαση σε ξένες αγορές. Τα μη εμπορικά εμπόδια πρέπει να μην υπάρχουν με κανέναν εμπορικό εταίρο πρέπει επίσης η Ευρώπη να μελετήσει και τα δικά της εμπορικά μέτρα για να δημιουργήσει μια πραγματικά ενιαία και ελεύθερη αγορά. Είναι καλό που βλέπουμε ε, την ίδια την Επίτροπο εδώ σήμερα, την κυρία ε, την κυρία, από το Λουξεμβούργο, την κυρία Λούλινγκ λέει κατά λάθο ο μιλητής και γελάει. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, αλλά πραγματικά είναι ένα προσωπικό ζήτημα που αφορά το πρόβλημα των δασμών για τα καύσιμα κατά την διαμεθοριακή μετακίνηση. Κυρία Ρέντινγκ, υπάρχει το θέμα των δασμών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να επιληθεί. Η Κομισιόν πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στα πλαίσια των θεμάτων που αντιμετωπίζει στον ΠΟΕ ε, με τις υφιστάμενες συμφωνίες για τα τεχνικά εμπόρια ε, ε, στο εμπόριο και τη συμφωνία TBT. Όσον αφορά τα FTA, πρέπει η συμφωνία αυτή να έχει επαρκή αμοιβαιότητα και πρόσβαση στην αγορά και στις δύο πλευρές, ώστε και να αυξηθεί η γνώση για τα μη δεσμολογικά εμπόρια, αλλά και να ξεκινήσει πόλεμος για την αντιμετώπιση τους. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ενημέρωση και στον ΠΟΕ και στον ΟΣΑ και σε όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για αυτά τα οποία έχουν γίνει γίνει αυτά τα οποία γίνονται και για πιθανή συσχέτιση της ύπαρξης μη θεσμολογικών εμπορίων και της, ε, ε, και της ύπαρξης και των μεριδίων αγοράς. Επίσης θα θέλαμε η Κομισιόν να αναπτύξει έναν ε, μηχανισμό έγκαιρο εντοπισμού αυτών των μη θεσμολογικών εμπορίων. Η έκθεση μας δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος με βασικούς εταίρους και τα θεσμικά όργανα για να μειωθούν τα δικαιολόγητα μη δεσμολογικά εμπόδια. Πρέπει να μελετηθούν ε, ιδιαίτερα τα LCD και τα SD γιατί στις αγορές αυτές υπάρχουν ευαισθησίες και να γίνει ε, ε, διάκριση μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων οικονομιών όπως είναι οι χώρες BRIC. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, των σκιωδών, τους σκιώδες ηγητές και όλους τους άλλους οι οποίοι συνδύασαν τις προσπάθειές τους σε αυτή τη σημαντική, την έκθεση που έγινε τόσο σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στάρντι. Και η φύση αυτής της συζήτησης και η σημασία της έχει σαν αποτέλεσμα να παρέμβουν ε, συνάδελφοι στο πλαίσιο της διαδικασίας του Catch the Eye. Ε, πρώτος είναι ο κύριος ε, Κασπάρη. Παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ρόμπερτ Στάρντι για την έκθεσή του, όπου πραγματικά μας δίνει μια πολύ καλή εποπτεία για όλες τις δυσκολίε που παραμένουν στο εμπόριο. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια συζήτηση στη Μήνη Ολομέλεια στις Βρυξέλλες ε, πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών ε, όσον και ε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί συζήτηση αυτή ο αρμόδιος επίτροπος. Ε, και εκφράσαμε την ε, ανησυχία ότι για αυτό τα περιεχόμενα τελικά της σύντησης αυτής δεν θα φτάσουν στην Επιτροπή. Και μου έκανε κατάπληξη όταν ε, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι η Κομισιόν δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι είναι μια, ένα θαυμάσιο παράδειγμα για ένα φραγμό στο εμπόριο και θεωρώ κύριε Επίτροπε ότι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό εφόσον λαμβάνετε σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όσον αφορά τους ε, φραγμούς ε, στην, ε, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, καθίστεται σαφές ότι ο μεγαλύτερος όγκος του εμπορίου τελικά λαμβάνει χώρα εκτός η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, βιομηχανικής της πολιτικής ε, αφο... Ε, βασίζεται στις πρώτες ύλε και τις σπάνιες γέες και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη κερδοσκοπία στην αγορά των πρώτων υλών. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις χώρες Μερκοσούρ και την Ινδία, έστω και αν στην Ινδία οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί τέσσερις φορές και η Ινδία ε, ε, συγγνώμη, δημιουργεί όλο και περισσότερους φραγμούς ε, στο εξωτερικό εμπόριο. Οι υπόλοιπε χώρες BRIC ξέρουμε ότι παίρνουν δασμολογικά μέτρα πολύ αρνητικά ε, κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εμπορική τους ε, πολιτική ε, και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και σημαντικοί περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Στάρντι ότι το ευρύ φάσμα ε, μεμονωμένων ε, μέτρων ε, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Θεωρώ ότι θα πρέπει σε συνολικό επίπεδο να βρεθούν απλές και απλά και ολοκληρωμένα μέτρα, ας πούμε προστασία της υγείας. Επίσης, πολύ συχνά βλέπουμε ότι λαμβάνονται μέτρα τα οποία στην ουσία είναι μέτρα προστατευτισμού και αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει και είναι προς το συμφέρον τους ε, να άρουν ε, τη, όλα, όλους τους μη δεσμολογικούς ε, φραγμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα, ο κύριος Τζέκετη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Στόρντι. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την έκθεση. Αλλά ούτε από πολιτική ούτε από οικονομική άποψη δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την έκθεση. Γιατί η μη δεσμολογική ε, φραγμή είναι απολύτω κατανοητή, γιατί υπάρχει μια χρηματοπιστωτική κρίση και διάφορε χώρε θέλουν να προστατεύσουν την οικονομία του. Το ελεύθερο εμπόριο ε, έφερε τις ε, χώρες αυτή την κατάσταση σε διάφορες αγορές. Όλοι έγιναν φτωχότεροι. Ε, η ανεργία έχει αυξηθεί. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να προωθούμε την ελεύθερη οικονομία, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε πατριωτικά ισχυρές οικονομίες. Γιατί ε, αυτό χρειάζεται χώρες που βρίσκονται σε μια συμμαχία μεταξύ τους και μπορούν να επικεντρωθούν στις τοπικές αγορές δημιουργώντας μια νέα βάση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφο, κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Στέρντι για τη δουλειά που έκανε και για τις προτάσεις του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προβλήματα στην Ευρωζώνη και τα το μέλλον μας όσον αφορά τον ανταγωνισμό μας σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ε, τίθεται εν κινδύνο. Πρέπει να φροντίσουμε όλα όσα γίνονται στον χώρο του εμπορίου θα γίνονται με δίκαιο και οικονομικά σωστό τρόπο για να μην βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση και όλα αυτά τα εμπόδια πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί στην ουσία πρόκειται για προστατευτισμό και αυτό δεν χρειάζεται στη σύγχρονη εποχή. Επίση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε ε, ε, τέτοιου είδους εμπόδια ότι οι συμφωνίες FTA θα είναι αποφελείς για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Γιατί θεωρώ ότι στο παρελθόν δεν έχουμε φροντίσει να το κάνουμε. Ε, Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζο Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για έναν ύμνο εδώ στο ελεύθερο εμπόριο. Ε, κάτι που ακούμε πολύ συχνά σε αυτούς τους ιερούς χώρους. Εδώ πρόκειται για, τους, ε, για, εμπορικού, για εμπορικούς φραγμούς που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην σημαίνονται καμία πρόοδος, έτσι λέγεται, αλλά τα πράγματα έχουν εντελώς διαφορετικά. Η απελευθέρωση και απορρίθμιση του διεθνούς εμπορίου οδήγησε στο κοινωνικό ντάμπινγκ καθώς και στο περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και δεν είναι το να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να υποτιμάται η εργατική δύναμη για να το εκφράσω έτσι και αυτό οδηγεί σε ακόμα περισσότερες δυσκολίες και τώρα για να αρθούν ορισμένοι φραγμοί ε, τελικά ε, θίγονται και κάποια μέτρα της κοινή ωφέλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δούμε, να εξετάσουμε ποιος είναι ο ρόλος του ελεύθερου εμπορίου. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχει ένα επιπλέον όφελος, όχι να ωφελεί τον ανταγωνισμό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κυρία Επίτροπε, καταρχήν θερμά συγχαρητήρια προς τον κύριο Στέρντι για αυτή την ε, πολύ σημαντική έκθεση η οποία ήρθε στο σωστό χρόνο και πραγματικά θα πρέπει να υποστηριχθεί από μέρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε οι μη δεσμολογικοί ε, φραγμοί να μειωθούν ούτως ώστε να γίνουν εφικτές οι, επενδύσεις στο εξωτερικό ε, στο άρθρο 206 της Σύνδεξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι σταδιακά θα πρέπει να καταργηθούν οι εμπορικοί φραγμοί και όσον αφορά τους μη δασμολογικούς φραγμούς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με, την, ε, με τα ζητήματα της εργασίας. Έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους που έχουν αυτούς τους μη θασμολογικούς φραγμούς όπως είναι η Ρωσία, η, η Κίνα και όλα αυτά περιορίζουν τις δυνατότητές μας σε αυτές τις αγορές και αντιβαίνουν στις προσπάθειες ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ελένα Μπασέσκου. Τα μη δασμολογικά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών παραγωγών και εξαγωγέων ε, σε ξένες αγορές είναι απαραίτητο. Θα πρέπει τα διεθνή πρότυπα να εφαρμόζονται σωστά. Η αμοιβαία πρόσβαση των αγορών και των δύο πλευρών ως μέρος μιας διμερούς συμφωνίας είναι απαραίτητο στοιχείο. Είμαι υπέρ της πρόθεσης ε, μιας, ε, ενός κώδικα, κωδίκων διοντολογίας της δημοκρατικές προμήθειας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες κρατικών προμηθειών τρίτων χωρών υπό δίκαιες και σωστές συνθήκες, ενώ θα πρέπει να δημιουργείται ένα σταθερό περιβάλλον ε, για τους Ευρωπαίους επενδυτές στο εξωτερικό. Υπογραμμίζω ότι είναι απαραίτητο να καταργηθούν οι περιορισμοί για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ένωση είναι σημαντικός εξαγωγέας υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Θα τελειώσουμε αυτό το σημείο με την παρέμβαση της κυρίας Επιτρόπου και Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, της κυρίας Ρέντινγκ, η οποία θα απαντήσει στις ε, παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ίντε και κυρίως ε, τον εισηγητή, τον Ρόμπερτ Στέρντι που ανέλαβε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα των εμπορικών φραγμών και κυρίως των μη δασμολογικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις αγορές τρίτων χωρών. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Επιτροπή το έχει επισημάνει αυτό στην πρώτη ετήσια έκθεσή της για τα εμπόδια στις επενδύσεις και το εμπόριο το Μάρτιο φέτος και η έκθεση ε, πηγαίνει ακριβώς στην καρδιά της πολιτικής μας για την εφαρμογή αυτών των θεμάτων. Η έκθεσή σας ενισχύει την πολιτική διάσταση ε, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε σημειώσει τις προτάσεις σας και όταν λέω έχουμε αναφέρομαι και εκ μιλάω και εκ μέρους του συναδέλφου Κάρτε Γκούχτ που είναι ο υπεύθυνος επίτροπος για το θέμα αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει την απομάκρυνση των ε, μη δίκαιων ε, μη δασμολογικών φραγμών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά με τους εμπορικούς μας εταίρους. Ε, θα κάνουμε απολύτως σεβαστό το δικαίωμα των εταίρων μας να θεσπίσουν ένα ε, δικό τους επίπεδο ε, προστασίας δημόσιας πολιτικής στον τομέα της υγείας, ε, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Ένα παράδειγμα ρυθμιστικής συνεργασίας όπου πρέπει να σας πω ότι και η Κομισιόν την προηγούμενη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου του 2011 ενημέρωσε το κοινοβούλιο για την, για στο, σε σχέση με την Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο στη Ουάσιγκτον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους ρυθμιστικούς τομείς η νανοτεχνολογία ας πούμε η, η, τεχνολογία πληροφορικής και υπολογιστών ε, ε, όσον αφορά το θέμα του, του Αμερικανικού Jobs Act παρακολουθούμε την νομοθεσία αυτή πολύ προσεκτικά και θα γνωρίζετε ότι κάποια από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία ευτυχώς δεν εγκρίθηκαν από την νομοθετική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης χρησιμοποιούμε τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μας για να αντιμετωπίσουμε τα ρυθμιστικά εμπόδια. Η συμφωνία με την Κορέα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για τέτοιε προσέγγισης γιατί συμπεριλαμβάνει εκτεταμένους κανόνες για διάφορα κλαδικά ρυθμιστικά ζητήματα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, ιατρικές συσκευές. Στην πρόσφατη συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής Εμπορίου που ε, συνήφθη υπό τη συμφωνία αυτή, ο Υπουργός της Κορέας και ο Επίτροπός μας κατάφεραν να σημειώσουν σημαντική προόδο για κάποια από τα εκρεμή ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούσαν τα αυτοκίνητα. Η σημασία των ρυθμιστικών ζητημάτων και η αλληλεπίδραση μεταξύ ε, των ανοιγμάτων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά θα συζητηθεί στην υψηλό επίπεδο συνάντηση που οργανώνει η Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Έχουμε σημειώσει τις προτάσεις σας για τις κρατικές προμήθειες, τις επενδύσεις, τις περιορισμούς των εξαγωγών. Θέματα που πράγματι είναι πολύ σημαντικά ε, στην εμπορική πολιτική του 21ου αιώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η απομάκρυνση των εμπορικών εμφραγμών είναι και παραμένει προτεραιότητα της εμπορικής μας πολιτικής επόμενη έκθεση για τα εμπορικά εμπόδια και τα εμπόδια στις επενδύσεις της Κομισιόν θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2012 και θα περιλαμβάνει και τις δικές σας προτάσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κύριε εισηγητά που βρίσκεται σε αυτή η έκθεση θα αποτελέσει έμπνευση και θα στηρίξει τη συλλογική δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Κρατών Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Με την ε, παρέμβαση της κυρίας ε, Ρέντινγκ Κλείνουμε τη συζήτηση. Θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Στόρντι και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ψηφίσουμε αύριο ε, το μεσημέρι στις 12. Κυρίες και κύριοι, η προσεχή συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο, 3η ε, 13 Δεκεμβρίου, από τις 9 ω τι 2 και από τις 3 ως τις 8 και στη συνέχεια από τις 9 ως τις 12 το βράδυ. Η εμερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας και σας εύχομαι καλή νύχτα.